τα διδάγματα τα οποία μπορούν να αντληθούν. Έχει το λόγο εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές φορές αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι ένα παράδειγμα ότι τα κοινοβούλια των κρατών μελών θέλουν και αυτά να κάνουν το ίδιο. of Οι ακροάσεις των Επιτρόπων πριν πάρουμε απόφαση σχετικά με την ψήφο εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Φανταστείτε, πριν αναλάβει το ρόλο της μια κυβέρνηση σε μια χώρα, κάθε υπουργός να περνάει από ένα εξαντλητικό έλεγχο για τρεις ολόκληρες ώρες πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιό του. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε. Πρέπει λοιπόν, και αυτό κάνει η έκθεσή μου, να προσπαθήσουμε ε, να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή με τρεις τρόπους. Πρώτον, ε, οι ερωτήσεις, το ερωτηματολόγιο η διερευνητική στόχη αυτού του ερωτηματολογίου. 42 ε, ερωτήσεις, 42 απαντήσεις. Εγώ προτείνω να μειωθεί ο αριθμός αυτός σε 25 ερωτήσεις, αλλά να μπορεί αυτός ο οποίος θέτει το ερώτημα να δευτερολογήσει μετά την απάντηση. Αυτό νομίζω θα επιτρέψει μια μεγαλύτερη διαδραστικότητα. Το θέμα δεν είναι να δώσουμε τον, τον λόγο στον μέγιστο αριθμό των βουλευτών, το θέμα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε τις περισσότερες πληροφορίες από τον υποψήφιο. Η δεύτερη πρόταση είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, θα αξιολογήσουμε τον υποψήφιο επίτροπο. Ε, τώρα ε, οι κανόνες μας δεν είναι ξεκάθαροι, ο κανονισμός μας. Οι συντονιστές συναντώνται και συζητούν και θα μπορούσε να ερμηνευθούν οι κανόνες μας να υπάρχει μία ψηφοφορία έτσι κι αλλιώς μετά από κάθε ακρόαση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο νομικά βέβαια είναι ισχυρό είναι η ψήφος του Κοινοβουλίου για το σύνολο της Επιτροπής. Οι μεμονωμένες επιτροπές και η ψήφος των μεμονωμένων επιτροπών, μεμονωμένων συγγνώμη επιτροπών δεν έχει νομικό βάρος παρόλα αυτά έχει πολιτικό βάρος. Με άλλα λόγια, μία ψηφοφορία για έναν επίτροπο θα πρέπει να γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αμφιβολίας και όχι σαν ρουτίνα. Και αν υπάρχει αρνητική φυσικά άποψη, αυτό έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεσή μου προτείνει να διευκρινίσουμε τις διαδικασίες αυτές. Ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θέλω να θέσω είναι το θέμα της ισορροπίας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμένει στην βελτίωση της ισορροπίας των φύλων. Παρ' όλα αυτά δεσμευόμεθα από τις προτάσεις ορισμούς που γίνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ε, πέρυσι τουλάχιστον μια χώρα πρότεινε δύο πρόσωπα και άφησε τον πρόεδρο της Επιτροπής να επιλέγει. Δηλαδή να το θεσμοποιήσουμε προτείνω αυτό. Κάθε χώρα, κάθε κυβέρνηση να προτείνει δύο επιτρόπους, ένα από κάθε φύλλο, στους οποίους έχει πλήρη εμπιστοσύνη η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι σε καλύτερη θέση να αποκαταστήσει την ισορροπία των φύλων του συνόλου της ομάδας και αυτό θα βελτιώσει κατά πολύ την κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις σε αυτή την έκθεση, αλλά αυτές είναι οι τρεις βασικές. Διαβάστε συνάδελφοι και τις υπόλοιπες γιατί βελτιώνουν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε μονάχα τη διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τότε που έχω γίνει βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντυπωσιάζομαι πάντα από το θέμα αυτό. Γιατί κατά την άποψή μου το σύστημα του διορισμού των επιτρόπων δεν ήταν ιδιαίτερα σαφές. Πρέπει να γίνουν λοιπόν τα απαραίτητα με τέτοιο τρόπο ώστε ο πρόεδρος μιας επιτροπής που κάνει ακρόαση επιτρόπου να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την καλύτερη επιλογή για τον επίτροπο. Όταν μιλάμε για επιτρόπους από μεμονωμένες χώρες, ούτε και αυτό το σύστημα είναι θετικό. Συμφωνώ μαζί σου, Ριχάρδε, ότι τα κράτη θα πρέπει να προτείνουν τουλάχιστον δύο υποψηφίους, αυτό θα ήταν πολύ καλό, λαμβάνοντας υπόψη και την εμπειρία των εμπειρογνωμών αυτών και το προφίλ γνώσεών τους, ώστε ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής να μπορεί να έχει μια πιο ε, εξισορροπημένη πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σφέρ Μπορσάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κόρμπετ και τους άλλους συναδέλφους από άλλες επιτροπές για το έργο που έχει γίνει στην έκθεση αυτή. Οι υποψήφοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή. Όταν θέλουμε να επιλέξουμε αυτούς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και το ηθικό ανάστημα των ανθρώπων αυτών αλλά και την εμπειρία τους στο αντικείμενο. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία θα πρέπει να εμπλέκει και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν περισσότερο στις ε, διαδικασίες ακρόασης. Προτείνω λοιπόν να υπάρχει και έλεγχος του βιογραφικού των υποψηφίων και υποστηρίζω την πρόταση να είναι δύο υποψήφοι ανά χώρα. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η διαδικασία της ακρόασης των επιτρόπων μια πολύ σημαντική διαδικασία διότι έτσι διαμορφώνεται ο δημοκρατικός έλεγχος μπορεί πραγματικά το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να ασκήσει τα δικαιώματά του και να δώσει όταν χρειαστεί την ψήφο εμπιστοσύνης συνολικά στην ίδια την κομισιόν. βεβαίως πρέπει να είναι μια διαδικασία πιο ανοιχτή στην ίδια την κοινωνία να μπορούν και οι πολίτες να συμμετέχουν και είχα την ευκαιρία όπως και εσείς να λάβω φέτος πέρυσι μάλλον μέρος σε αυτή τη διαδικασία και λάβαμε πολλά email από πολίτες που έθεταν ζητήματα για διάφορους commissioners οι οποίοι είχαν προταθεί. νομίζω ότι πρέπει ως βουλευτές να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο και να έχουμε και περισσότερο χρόνο να υποβάλουμε ερωτήσεις να μην αφήνουμε όλο το παιχνίδι μόνο στους συντονιστές τέλος θέλω να θέσω ένα βασικό ερώτημα στα ελάχιστα δευτερόλεπτα η επιτροπή πρέπει να είναι πραγματικά το ανεξάρτητο όργανο έτσι όπως τη θέλουμε και να μην υπηρετεί την τρόικα. αυτό είναι πολύ σημαντικό κύριε τίμερμανς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρία. Κύριος Άρνετ είναι ο τελευταίος κύριε Κόρμπερτ, Εγώ σέβομαι τις προσπάθειές σας να, κάνετε, να είναι πιο υπόλογη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια καλή πρόταση εδώ και έχουμε και γνωμοδοτήσει από άλλες επιτροπές. Είναι καλό το να έχουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά αν υπάρξει κάτι τέτοιο στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούμε ίσως επιτέλους να έχουμε μια πραγματική συζήτηση εδώ. Εμείς δεν βλέπουμε τον ελέφαντα όμως που είναι μέσα στην Ολομέλεια. Οι επίτροποι έχουν τεράστια εξουσία και μόνο μια, ένα υποψήφιο μπορούμε να ακούσουμε για ε, κάθε θέση. Μου θυμίζει κάποια άλλη ένωση που είχε μονάχα ένα υποψήφιο για κάθε θέση. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς δίνουμε στα άτομα αυτά τις τεράστιες αυτές εξουσίες και όχι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το να έχουμε μη εκλεγμένους επιτρόπους, έχουμε ε, επιτρόπους που δεν είναι υπόλογοι σε κανένα. Ευχαριστώ κύριε Άνοτ. Ο κύριος Τίμερ μας έχει το λόγο από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσους υποψηφίους ακούει στην Άνω και στην Κάτω Βουλή της χώρας του. Ας μην ξεκινήσω μια τέτοια συζήτηση τώρα βέβαια. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κόρμπετ, για μια εξαιρετική και ζυγισμένη πρόταση. Για ένα θέμα το οποίο όπω κατανοείται έχει πάρα πολύ μεγάλο βάρος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τον επιδιωκόμενο στόχο έτσι ώστε οι ακροάσεις να γίνονται πιο δυναμικές και ευέλικτες. Οι ακροάσεις αυτές δεν επιτρέπουν να συγκρίνονται οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά πόσον είναι συμβατές με τη συνθήκη, αλλά να ορίζουν και σωστά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ήμουν κάποτε υπουργό. μετά έγινα επίτροπος και ξαφνικά από πολιτικός έγινε ένας ανώνυμος ε, γραφειοκράτης και ο έλεγχος τον οποίο υπέστην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο σκληρός από τον αντίστοιχο έλεγχο στην άνοβουλή της Ολλανδίας. Λοιπόν, πόσες κυβερνήσεις, δεν ξέρω τώρα τον αριθμό, υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις στις οποίες οι υπουργοί δεν εκλέγονται. Λοιπόν, ε, βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα έχουν διαφορετική, υπάρχει διαφορετική πραγματικότητα από την εικόνα που έχουμε για αυτά. Θα πρέπει λοιπόν οι ακροάσεις να οργανώνονται με ανοιχτό τρόπο, με δίκαιο τρόπο και θα πρέπει να ακολουθείτε η διαδικασία των ερωτοαπαντήσεων και στην γραπτή φάση και στην προφορική φάση. για τους ε, υποψηφίους ε, αντιπροέδρους που έχουν οριζόντιες ευθύνες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε πολλαπλές κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει ίσως να υπάρχει μια ανοιχτή διάσκεψη των προέδρων γενικότερα η περίοδος αυτή έγκρισης θα πρέπει να κρατά τόσο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι μόλις λήξει η εντολή του προηγουμένου επιτρόπου θα ξεκινήσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο νεοεκλεγής επίτροπος. Έτσι θα γίνονται έγκαιρα και ζυγισμένα, σταθμισμένα οι επιλογές. Σχετικά με την οργάνωση τώρα των ακρόσεων ε, εμείς συμφωνούμε για την έξεση των γραπτών ερωτήσεων από 5 σε 7. Ε, επίσης θεωρούμε ότι είναι θετική η πρόταση για τον περιορισμό των προφορικών ερωτήσεων σε 25 ε, με δυνατότητα δεύτερης ερώτησης στη συνέχεια. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπέρ του στόχου του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη και διαφανής για τον Ευρωπαίο πολίτη η ακροαματική διαδικασία. Αλλά θα πρέπει βέβαια να μπορούν τα μέλη του Κοινοβουλίου να ελέγξουν σωστά τον υποψήφιο. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Είναι δικαίωμα λοιπόν των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα θέτουν τις ερωτήσεις αυτές στον υποψήφιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στη διάθεση του Κοινοβουλίου για την εξέταση θεμάτων όπως η σύγκρουση συμφερόντων των υποψηφίων επιτρόπων θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροπολογήσει τον κώδικα συμπεριφοράς τον οποίο ακολουθεί σύμφωνα και με τις απόψεις ε, του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει οι υποψήφοι επίτροποι να αξιολογούνται επί τη βάση των προσωπικών τους ικανοτήτων σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο και τη φύση του χαρτοφυλακίου και γι' αυτό θα πρέπει τα αποτελέσματα της ακροάσεως να δημοσιεύονται μεμονωμένα σε κάθε περίπτωση 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας. Σχετικά τώρα με τους αντιπροέδρους νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες του κάθε επιτρόπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξετάσει τις συγκεκριμένε προτάσεις που κάνατε όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ακροματική αυτή διαδικασία για την εξέταση των υποψηφίων. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ θερμά κύριε Κόρμπετ, εξ ονόματος όλης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τι μας. Ακόμα και αν ε, εσείς ε, θέλετε να απαντήσετε ίσως κύριε Κόμπετ. Ακριβώς ε, θέλησα να διατηρήσω ένα λεπτό από το χρόνο μιλίας που μου έχει δοθεί για να απαντήσω και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ένα πολύ ψηλό βαθμό συνένεση ανάμεσα στι πολιτικέ ομάδε για τι προτάσει που έκανα και χαίρομαι όμω πάρα πολύ που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιο ο κύριο Τίμερμαντ σχολίασε πολύ ευνοϊκά ορισμένα από τα πράγματα που δεν είχα το χρόνο εγώ να σχολιάσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας στηρίζει τόσο ένθερμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνεί από ό,τι φαίνεται με όλες τις ε, προτάσεις μας. Βέβαια πολλές φορές ξέρετε ότι ο διάβολος μπορεί να κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για άλλη μια φορά όμως σας ευχαριστώ ολόθερμα για την υποστήριξή σας και να σας ευχαριστήσω επίσης και για τα όσα είπατε στην προηγούμενη συζήτησή μας που νομίζω ότι πραγματικά δώσατε κάποια πολύ θετικά στοιχεία όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε συνάδελφε Κόρμετ. Συνάδελφε Κόρμετ, εξαιρετικά γνωρίζετε τον κανονισμό και πολύ κομψά προχωρήσατε με την εξάντληση των τεσσάρων λεπτών. Δεν είχατε περισσότερα λεπτά. Εν πάση περιπτώσει,